Αγαπητοί συνάδελφοι, Σα if ε, σας παρακαλώ, ας αρχίσουμε σιγά σιγά. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι το ιδεώδες πρόγραμμα, γιατί συνεδριάζει ολομέλεια ε, και έχει έρθει ο κ. Βαν αλλά τι να κάνουμε, αυτό το πρόγραμμα μας δώσανε. Και ας συνεχίσουμε. Το σημείο 10. Θέσπιση ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό. Η κυρία Γκέπχαρτ είναι συγγήτρια. Adopted to launch Το κοινοβούλιο εδώ θέλει ενισχυμένη συνεργασία στον ευαίσθητο αυτό το τομέα που αφορά το διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό και ε, ε, υπόψη σας ότι είναι πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκέπχαρτ, την εισηγήτρια και μετά αν θέλει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει τίποτα να προσθέσει. Για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψε. Παρακαλώ, πρώτα όμως η εισηγήτρια, κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όντως είναι καινοτομία αυτή. Ενισχυμένη συνεργασία χρησιμοποιούμε σε αυτό το τομέα για πρώτη φορά και θα γνωρίζετε και από την περασμένη θητεία ότι εγώ δεν είμαι και καμιά τεράστια ε, θαυμάστρια και υποστηρίκτρια αυτής της διαδικασίας γιατί ήταν μάλλον διακυβερνητικό το μέσο αυτής της συνεργασίας. Βέβαια, απέτυχε η πρώτη νομοθετική απόπειρα, διότι στο Συμβούλιο ακριβώς δεν υπάρχει δυνατότητα ομοφωνίας. Οι πολίτες μας όμως έχουν πάρα πολλά προβλήματα, άνδρες και γυναίκες, και πρέπει να λυθούν. Γι' αυτό είπαμε ότι εντάξει, ας το κάνουμε. Ο τότε επίτροπος ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικός, δεν ήθελε πάρα πολύ να το προωθήσει και μας έλεγε πάντα ότι ναι καλά, το ελέγξουμε, θα το δούμε. Ε, γι' αυτό χαίρομαι που η νέα επίτροπος η κυρία Ρέντινγκ αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία σε περίπτωση που νέα κράτη-μέλη, ε, ε, ε νέα κράτη-μέλη, συγγνώμη, το ζητήσουν. Το 1 τρίτο. Και στο μεταξύ δεν είναι νέα, αλλά 14 τα κράτη που το έχουν ζητήσει και θέλουν να συνεργαστούν και έχω την αίσθηση ότι θα αυξηθούν ε, ακόμα περισσότερο και είναι πολύ καλό. Ε, δεν είναι ένας πολύ στενός κύκλος λοιπόν ε, χωρών, αλλά πολύ περισσότερες από το 1 τρίτο που θέλουν να συμμετέχουν. Και αυτό είναι καλό. Και την περασμένη εβδομάδα τώρα η Ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία συμφώνησε και υπερψήφισε για την ενισχυμένη συνεργασία και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια καλή επίλυση του θέματος. Κάτι άλλο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν είμαστε πλέον αρμόδια ε, επί της ουσίας επιτροπή όπως την περασμένη θητεία έχουν ανατραπεί τα πράγματα ε, γιατί άλλαξε ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τώρα η νομική επιτροπή είναι εκείνη που κάνει την κύρια έκθεση και εμείς νομοδοτούμε. Την περασμένη φορά είχαμε κάποιες δυσκολίες στη συνεργασία γιατί ο συνσηγητής ήταν αρκετά συντηρητικός. Την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να συζητήσω και να συνεργαστώ με τον κύριο Σβίφκα ε, και είναι καλά τα νέα, είναι πολύ πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί μας και δεν το βλέπει τόσο στενά ε, όσο ο προκάτοχός του στη Γιούρη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Μπορούμε λοιπόν να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά και επίσης είχαμε και ανταλλαγέ απόψεων επί τη ουσία για τα θέματα αυτά που μας απασχολούν και πρέπει να συζητούμε. Κάτι άλλο που έχω να σας πω, βέβαια αυτό πρέπει να επαληθευτεί ακόμα, γιατί μιλάμε αγγλικά μεταξύ μα και δεν είναι μητρική γλώσσα, είναι τρίτη γλώσσα και εκείνον και για μένα, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί. Ε, Παρ' όλα αυτά, ελπίζω να μπορέσω να τα αποδώσω αυτά και να σας πω τι έγινε. Χρειαζόμαστε μια αλλαγή και μια οδηγία η οποία να είναι φιλική προς τους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε και συμφωνήσαμε με τον εισηγητή να μην έχουμε ένα shopping, δηλαδή να επιλέγει ο καθένας ό,τι θέλει, ε, να είναι σαφείς οι κανόνες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου θέλει ο ένας σύζυγος να χωρίσει αλλά ο άλλος όχι να υπάρχει ε, σαφής ιεραρχία και να μην επιλέγει ο ισχυρότερο σύζυγος με βάση ποιο δίκαιο θέλει να ζητήσει διαζύγιο, διότι το δίκαιο για το διαζύγιο στα κράτη-μέλη είναι πολύ διαφορετικό από χώρα σε χώρα για να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Τα δικαιώματα επιμέλειας στη Γερμανία, ας πούμε, λύνονται ταυτόχρονα με το διαζύγιο, ενώ στη Γαλλία είναι διαφορετικές διαδικασίες, τελείως διαφορετικές. Δηλαδή θα πρέπει να γνωρίσουν και τα δύο ε, μέρη και οι δύο σύζυγοι τι ισχύει και πώς θα κανονίζουν την πορεία τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης εκεί που υπάρχει δυνατότητα επιλογής, διότι συμφωνούν και οι δύο ε, να χωρίσουν, να είναι πολύ καλά ενημερωμένοι και να επιλέγουν με τα λόγου γνώσεως. Και χρειάζεται λοιπόν πολύ μεγάλη μελέτη, έρευνα και έλεγχος και θα το ζητήσω αυτό με τροπολογίες. Έχω την αίσθηση ότι και ο κύριος Βίφκα συμφωνεί μαζί μου και θέλει να πάρει αυτή την τράπο. Σας είπα ότι έχω ένα πρόβλημα εκεί. Δεν ξέρω, μπορεί να μας διαφωτίσει το Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για ποιο λόγο στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4 τα κάνετε αυτά. Στην περασμένη θητεία. Και πάλι επαναλαμβάνω σύμφωνα με ποιο δίκαιο και ποια δικαιοδοσία στο ΔΕΛΤΑ λέει το δίκαιο του κράτου στο δικαστήριο του οποίου προσφεύγει κανεί. χωρίς κανένα όρο και προϋπόθεση. Αυτό για να το καταλάβω. Τι σημαίνει στα 27 κράτη. Μπορεί οποιοδήποτε δικαστήριο, δηλαδή ή μόνο στα κράτη που συμμετέχουν σε αυτή την οδηγία. Μπορεί κάποιο να προσφύγει σε ένα δικαστήριο χωρίς να υπάρχει καμία προϋπόθεση και κανένα όρο. Φοβάμαι ότι αυτό είναι τώρα το shopping, ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε και διαλέξτε. Στην πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην πρώτη θητεία, αυτό ήταν μέσα και είπαμε ότι είναι επικίνδυνο και πάλι ξανά εμφανίζεται και το ίδιο στο άρθρο 4. Εάν οι δύο δεν συμφωνούν και πάλι στο Δέλτα λέει και προβλέπεται το κράτος, το δίκαιο του κράτους στο δικαστήριο του οποίου έχει προσφύγει κανείς. Και πάλι αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εάν δεν ισχύουν τα τρία προηγούμενα α, β, γ, ε, βρίσκει εφαρμογή το δέλτα. Γι' αυτό δεν θέλω να είναι τόσο ανοιχτά όλα και τόσες πολλές οι δυνατότητες. Αλλιώς δεν μπορώ να το δεχτώ. Κάτι άλλο που βρίσκω πολύ ωραίο στο άρθρο 7 γίνεται λόγος για τη δημόσια τάξη, order public. Το είχαμε προτείνει αυτό, στην πρώτη εκδοχή δεν το είχε μέσα. Μερικά από αυτά που ζητήσαμε εμεί στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου επανέρχονται στην πρόταση και χαιρόμαστε γι' αυτό και ε, μπορούμε να πούμε ήδη ότι έχουμε επηρεάσει τι καταστάσει ω Κοινοβούλιο. Βεβαίω δεν έχουν λήξει τα πάντα. Εγώ περίπου το βλέπω αυτό τώρα ως δεύτερη ανάγνωση. Γιατί ε, στην περασμένη θητεία και πάλι στο Κοινοβούλιο είχαμε πολύ μεγάλη πλειοψηφία για τη δική μας θέση και θα χρησιμοποιήσω ως βάση για την εργασία μου και για τις προτάσεις μου αυτή την απόφαση του Κοινοβουλίου. Και αν συμφωνείτε, θα προχωρήσουμε έτσι όπως σας προτείνω. Ο εισηγητής μου είπε ότι θέλει να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Βεβαίως θα πρέπει να συμφωνήσουν και τα μέλη της Επιτροπής μας. Ε, υπάρχει λοιπόν η νομική βάση για να βρούμε μια λύση για τους πολίτες μας, άνδρες και γυναίκες. Ελπίζω να προσθεθούν και άλλα κράτη-μέλη και κάποια στιγμή και κράτη τύπου Σουηδίας και άλλα να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί στο κάτω-κάτω πρόκειται για τα δικαιώματα των δικών τους πολιτών και γι' αυτούς ενδιαφερόμαστε. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αλλάξουμε ε, την κείμενη νομοθεσία και το δίκαιο των κρατών μελών. Αλίμονο, δεν έχουμε τέτοιε εξουσίε βάσει των συνθηκών εμεί. Αυτό που θέλουμε είναι να βοηθούμε του πολίτες να τους διευκολύνουμε τη ζωή και το διαζύγιο. Έτσι ώστε τα αρμόδια δικαστήρια να επιλαμβάνονται και να εφορμάζεται το εκάστοτε δίκαιο όπως πρέπει και όχι και κλεισμένο των θυρών ή ε, να, βρίσκουν κλειστές μάλλον τις πόρτες στο δικαστήριο όταν θέλουν κάποιοι να προσφύγουν σε αυτά. Γιατί μπορεί κάποια ζευγάρια να έχουν παντρευτεί με βάση κάποια νομοθεσία, στο μεταξύ να ζουν σε άλλο κράτος και να ε, υπάρχει πρόβλημα... Αυτά εισαγωγικά θα προσπαθήσω να δουλέψω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Η γραμματεία μου είπε ότι το σχέδιο γνωμοδότησης θα πρέπει να είναι στις 27 Σεπτεμβρίου και θα ψηφιστεί. Ναι. Και θα προσπαθήσουμε το συντομότερο να προχωρήσουμε για να βρούμε μια ρύθμιση που να εξυπηρετεί ε, και να βοηθάει τους πολίτες και να έχει νόημα και να είναι όσο γίνεται πιο ανοιχτή για να μην ε, αποκλείει κανένα. Βλέπω και την κυρία Βέλτ, η οποία ήταν σκιώδη συγγήτριά μου. Ε, και υπάρχουν ειδικά προβλήματα, α πούμε, στη χώρα τη επιτρέπονται γάμοι ομοφυλοφίλων, σε άλλα κράτη ε, όχι. Θα πρέπει να λυθούν και αυτά τα προβλήματα. Και ε, είναι θετική νομίζω η αφετηρία και μπορούμε να συνεργαστούμε για να τη βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ, όλοι, ο Πρόεδρος, στα γερμανικά. Και τώρα θα ακούσουμε την κομισιόν, τους, τους εκπροσώπους της Mrs. Mr. Zalewski, Ο κύριος Ζαλεύσκη ή η κυρία Σασταμόνεν. Έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω με ευχαριστίες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι ενήργησε με τόση ταχύτητα και αποτελεσματικότητα και έδωσε το πράσινο φως στην αρχική μας πρόταση για αναβαθμισμένη συνεργασία εν ώψη λήψης αποφάσεως το οποίο αποδεικνύει ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Και αυτό παρά το ότι μόνο κάποια συγκεκριμένα κράτη, μια ομάδα των κρατών στο Συμβούλιο έδειξε τον δρόμο για το μέλλον όσον αφορά αυτό το λεπτό θέμα του διαζυγίου και όσον αφορά το εφαρμοστείο δίκαιο εις περιπτώσεις τέτοιων διαφορών. Επίση, uh, Επίσης, δεν μπορώ να συμφωνήσω με την συγκεντρία ότι πρόκειται για μια ανοιχτή ενισχυμένη συνεργασία. Οπότε, να έχουμε περισσότερες χώρες οι οποίες να μπουν στο χώρο πέραν αυτών που ήδη έχουν ε, προσχωρήσει γιατί πήγαμε στο 9 και πήγαμε στο 14 ε, όσον αφορά τον αριθμό εκείνων που προσυπέραψαν εκείνο το κείμενο, το κείμενο εκείνο το οποίο πέρασε εδώ στο Κοινοβούλιο οπότε και γι' αυτό ελπίζουμε ότι και άλλοι πρόκειται να προσχωρήσουν σε αυτή την ε, πρωτοβουλία και τώρα αυτό το οποίο θα υπάρχει ο συνέπειο ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κείμενο γιατί έχουμε εδώ αυτές τις διατάξεις που προτείνουν θεσπιστούν για τους πολίτες της Ένωσης όσον αφορά αυτόν τον κανονισμό του οποίου αφετηρία είναι για μας η πρόταση όπως ε, διατυπώθηκε ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο κοινοβούλιο πρόσφατα γιατί πραγματικά ισχύει ότι προσπαθούμε να καλύψουμε και να λάβουμε υπόψη τα όσα είπε το Κοινοβούλιο στην προηγουμένη θητεία. Και αυτά όντω έχουν καλυφθεί από το κείμενο. Γενικώ αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα. Αυτό σημαίνει επίση ότι το κριτήριο για το εφαρμοστείο δίκαιο θα πρέπει να είναι τέτοιο που να είναι η, η ένωμη τάξη εκείνη που είναι πιο κοντά στο ζεύγος. Οπότε ξεκινούμε με το πρώτο κριτήριο το, που είναι η συνήθις κατοικία. Βέβαια σε περίπτωση που δεν έχουν διαλέξει το χρώμα στο δίκαιο τα, τα, τα, τα, δύο μέρη, δηλαδή, το, ζευγάρι. Τώρα όσον αφορά το φαρμαστείο δίκαιο θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν κάποιες σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες θα ορίζεται φαρμαστικό δυνάμει του άρθρου 4. Αυτό είναι η τελευταία περίπτωση κατά σειρά τελευταίο κριτήριο κατά σειρά εφαρμογής, γιατί αυτό σπανίως εφαρμόζεται στην πράξη ε, δεύτερος τόσο του δονισμού είναι το να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Διότι τώρα θα έχουμε την περιορισμένη αυτονομία του διαδίκου. Οπότε οι διάδικοι μπορούν να διαλέξουν το ορμοστήριο. Όταν υπάρχει μια τέτοια οικογενειακή διαφορά. Η προηγουμένη συμφωνία θα καλύπτει και τα συνετικά διαζύγια. Επίσης, θα δούμε το πρώτο θα γίνει με την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Οπότε να καλυφθούν αυτά τα τέσσερα σημεία και το θέμα του εφαρμοστικού δικαίου. Αυτό δεν που θέλουμε να σας τονίσουμε είναι το ότι lex φορεί σημαίνει το εφαρμοστικό δικαίου. Αυτό δηλαδή που καλείται να εφαρμόσει το δικαστήριο. Το θέμα είναι η δοσηδικία πώς θα κανονιστεί, ποιο θα είναι το δικαστήριο που θα επιληφθεί. Έχουμε επίσης και τον κανονισμό Βρυξέλλες Α, Βρυξέλλες Β. Στα λατινικά δηλαδή, εκεί ορίζονται τα θέματα που αφορούν τη δοσηδικία, ποιο είναι το δικαστήριο που θα επιληφθεί. Οπότε, στη συνέχεια θα δούμε ότι το δικαστήριο θα πρέπει να εφαρμόσει αυτό το οποίο προβλέπεται από, αυτή την ε, προ, προκείμενη ρύθμιση. Επομένως έχουμε από αυτούς, τους δύο τρόπους τον καθορισμό του οποίου θα είναι το δικαστήριο και έτσι δεν είναι δυνατόν να έχουμε την περίπτωση του να επιβάλλει ένας από τους δύο το εφαρμοστείο δίκαιο ή το δικαστήριο που θα επιληφθεί. Οπότε, ακριβώς και εμείς αυτό θέλαμε, το να, αποφύγει κάποιος ε, την ε, του το να επισπεύσει την, ε, την αίτηση διαζυγίου ήταν και αυτό ένας από τους λόγους που κάνουμε αυτό το σχέδιο κανονισμού. Άρα θέλουμε να είναι αντικειμενικά τα κριτήρια αυτή η σύνδεσμη, η συνάφεια τέλο πάντων του, του, του, των διαδίκων με το εφαρμοστικό δίκαιο. Επίσης, σε αντίθεση με το σχέδιο κανονισμού του 2006, ναι. αυτό το νέο σχέδιο κανονισμού δεν περιέχει ρυθμίσει σχετικά με την ένομη τάξη. Γιατί, τώρα βρισκόμαστε σε ενισχυμένη συνεργασία η οποία ενισχυμένη συνεργασία αφορά μόνο αρμοδιότητες της Ένωσης. Γιατί έχουμε εδώ ένα δεδομένο, ένα κεκτημένο το οποίο καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη και επομένως αυτά τα θέματα, τα θέματα της ένομης τάξης καλύπτονται από την προηγούμενη ρύθμιση. Επομένως τώρα έχουμε ένα καινούργιο νομοθέτημα το οποίο είναι αυτάρκες, αυτόνομο κατά κάποιο τρόπο, αυτοτελές. Και έχουμε αυτά τα επιπλέον περισσότερα δηλαδή άρθρα στο νέα πρόταση της Κομισιόν που είναι πολύ παραπάνω από τα, τις προηγούμενες πρότασεις. Φυσικά ε, παρακολουθήσαμε και λάβαμε υπόψη τα όσα προέκυψαν την προηγούμενη διαπραγμάτευση. Επίσης, το Κοινοβούλιο και η συγκεκριμένη Επιτροπή σα προτίθεστε να διεκπαιρεώσουμε ταχαίω το θέμα αυτό. Οπότε και είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι εκκρεμεί πολύ καιρό αυτό το θέμα από τότε που ξεκίνησε η πρώτη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει η νομοπαρασκευαστική διαδικασία με μεγάλη προσοχή, ιδίω σε όσο αυτά που μα είπε η εισηγήτρια, γιατί θα πρέπει σε όσα σημεία υπάρχει πρόβλημα να ζητηθούν κάποιε λύσει που θα είναι δόκιμες, θα εξυπηρετήσουν του Ευρωπαίους. Και αυτό να γίνει σε εύλογο χρόνο, μη χρονίσει. Και πάλι ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για τα όσα κάνατε μέχρι τώρα και βεβαίω και προτιθέμεθα να συνεργαστούμε ευχαριστώ μαζί σα στη συνέχεια. Thank you. Ευχαριστούμε, κυρία Σαταμόινεν. Λοιπόν, τώρα έχουμε λίγη ώρα για συζήτηση. Η κυρία Ιντφελτ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια. Είναι καλό να εργαστούμε ε, γρήγορα. Έχω δύο ερωτηματικά εγώ. Διερωτώ με, γιατί είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε και τη διαδικασία αυτή. Τι γίνεται. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο έτσι ώστε να μπορούν όταν ενταχθούν και νέες χώρες σε αυτή τη διαδικασία να είναι όλα εντάξει. Δηλαδή να μην είναι όλα πάρα πολύ προσιλωμένα και στατικά στο τι συμβαίνει στα 14 κράτη και άμα έρθει και άλλη μια χώρα να μην μπορούμε να το προσαρμόσουμε. Ε, επίσης, ακούω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλάει για μια φυγή ορμητική προς τα δικαστήρια, rush to court. Δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένο αυτό. Καμιά φορά ε, θα πρέπει ε, να ξέρουμε ότι είναι ε, και προς όφελος και του ασθενέστερου συζύγου να ε, βγει το διαζύγιο με το σωστό τρόπο ε, να είναι η διαδικασία καλή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Ρομέρο Λόπες. Θα ήθελα μερικές παραπάνω πληροφορίες όσον αφορά τον ελλογοκρανισμό γιατί κάτι δεν κατάλαβα καλά από τη συζήτηση. Τι γίνεται όσον αφορά τους διαμένοντες στην Ευρώπη υπηκόους τρίτης χώρας. Ή ανάποδα, οι ε, Ευρωπαίοι υπήκοοι που παντρεύονται κάποιον από τρίτη χώρα και διαμένουν εδώ. Τι γίνεται, θα ισχύσει το άρθρο 4 και το άρθρο 3 προϋποθέτει αμοιβαία συμφωνία, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι, κυρίως όσον αφορά τις γυναίκες, συνήθως στις τρίτες χώρες υπάρχει διεθνής διάκριση. Οπότε θα έπρεπε να ισχύσει το άρθρο 4 και να μπορούν να αποφασίσουν όπως προβλέπει εδώ δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μόνιμης κατοικίας. Και αυτό θα ήταν πρόοδος ουσιαστική όσον αφορά την ένταξη των εν λόγω προσώπων. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα If there is a perspective already now that more member states... Τι γίνεται. Ε, που τώρα θα διευρυνθεί κύκλος των συμμετοχών των κρατών μελών. Τι, θα γίνει, τι εξελίξεις προβλέπονται, λέει η κυρία Κέλλαρ και Όσο επιτοπλίστων συμφωνώ με όσα είπατε κυρία εισηγήτρια. Συμφωνώ. Τώρα για κάτι άλλο. Αν κατάλαβα καλά, αυτή η ενισχυμένη συνεργασία δεν καλύπτει τα θέματα ε, κυριότητος, το τάτα ε, ε, εμπράγμα της ιερτησίας. Πώς το ρυθμιστούν αυτά, θέμα της περιουσίας δηλαδή. Νομίζω υπάρχει αυτή η διαδικασία η οποία προβλέπεται αλλά η οποία είναι πάρα πολύ μακρά. Οπότε, σε περίπτωση που είναι κάποιοι που έχουν πρόβλημα που μειονεκτούν, θα πρέπει κάτι να ρυθμιστεί. Πρόεδρος, ε, αν δεν θέλουν να συναντηθεί το λόγο, τότε να μας απαντήσει η Κομισιόν σε σχέση με αυτά που ρωτήσαμε, αλλά πρώτα να είδε το λόγο η Η Κομισιόν πρώτα, η Κομισιόν. Ναι, Πρόεδρε. Δεν θα με γρηγορήσω. Ρωτήθηκε αν υπάρχουν και κάποια άλλα κράτη-μέλη... ή στο Συμβούλιο από τότε που από τότε που έγινε αυτή η συμφωνία, όχι από, τι 14, από τα 14 κατημέλη τα οποία συμφωνήσαν δεν είχαμε και άλλε εξελίξει. Είπαμε απλώ ότι πιστεύουμε, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προσχωρήσουν κι άλλοι και θα έρθουν στην ώρα του. Μόλι έρθει η ώρα τη απόφαση για την ε, ενισχυμένη συνεργασία, με την ενισχυμένη συνεργασία, οπότε τότε θα έχουμε και άλλε αιτήσει ε, Οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να πάρει τι αποφάσεις που πρέπει. Μόλις αυτές οι χώρες έχουν μπει στο χώρο τώρα όσον αφορά τα περιουσιακά. Ε, αυτό το σχέδιο εγγονισμού αφορά τα μη περιουσιακά θέματα. Βέβαια, εμείς επεξεργαζόμαστε κάποιο κείμενο όσον αφορά τις συνέπειες επί της περιουσίας συνέπειε από τη σύναψη γάμου και κατόπιν από το διαζύγιο. Βέβαια. Οπότε, σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να επιληθεί η σύγκρουση αντιφατικών κανόνων δικαίου. Όμως θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται όσον αφορά το εφαρμοστείο δίκαιο για τη διατροφή. Οπότε πρέπει εμείς τελικά να βρούμε κάποια λύση που να είναι συνεπής με το όλο πλέγμα κανόνα δικαίου που θα ισχύουν. Νομίζω εκάλυψα τις ε, ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Back to you, Mrs. Ωραία, κυρία Γκέμπχαρτ τώρα πάλι. Ε, ευχαριστώ. Τώρα αυτά που είπατε με κάνουν να θέλω να μιλήσω με την ώρα. Πόσο σημαντικό να έχουμε ένα ευρωπαϊκό οικογενειακό κώδικα που θα ήταν πραγματικά το σκοπιμότερο και το καταλληλότερο γιατί Έχουμε μεμονωμένα ε, ζητήματα, θέματα επιμέλειας, είπαμε διατροφής, ε, θέματα περιουσιακά και πάει λέγοντας. Είναι πολλά τα ζητήματα που τίθενται σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό. Δεν ρυθμίζονται καθόλου όλα αυτά, ούτε μπορούν να ρυθμιστούν άλλωστε. Εδώ πρόκειται μόνο για τη διαδικασία. Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο, ποιο δικαστήριο επιλέγεται για να αποφαίνεται και βάσει ποιου δικαίου εκδίδεται το διαζύγιο. Όλα τα υπόλοιπα δεν καλύπτονται αυτά. Ας πούμε, ζητήματα περιουσιακά, στα οποία αναφερθήκατε κυρία Χέλερ, ακόμα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή λύση και είναι πολύ σημαντικό ακριβώς να είναι ενήμερη η συνένεση με τα λόγου γνώσεως εκείνοι οι σύζυγοι που γνωρίζουν ότι ζητούν διαζύγιο βάση συγκεκριμένη νομοθεσία να ξέρουν ακριβώ και οι δύο τι συνέπειες θα έχει αυτό και ε, πώς θα λυθούν αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό λέμε να είναι ενημερωμένοι. Το ίδιο ισχύει για θέματα επιμέλειας, για θέματα διατροφή, Βρυξέλλες 2α όπως είπαμε ε, προηγουμένως. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γι' αυτό μου λείπει στην πρόταση κανονισμού αυτό το στοιχείο και θέλω να, να μπει για να ξέρει ο κόσμος ακριβώς. Αυτή η ενημέρωση για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν κάποιος επιλέγει μία χώρα βάσει της ε, νομοθεσίας της να χωρίσει, να ξέρει ακριβώς τι σημαίνει συγκεκριμένα αυτό. Ε, πάρα πολύ σημαντικό. Και συμφωνώ απολύτως. Τώρα, από εκεί και πέρα, κυρία Ρομέρο, με ρωτήσατε τι γίνεται με θέματα ένταξης ε, και σωμάτων στην κοινωνία, δεν μπορώ να τα απαντήσω αυτή τη στιγμή. Να το ελέγξω και θα σας πω, θα το κοιτάξω και θα σας ενημερώσω. Και τι γίνεται με τις πολίτε τρίτων κρατών, θα σημείωσα τα ερωτήματά σας και στο σχέδιο έκθεσης θα τα συμπεριλάβω για να δούμε ακριβώς πώς θα βρούμε μια λύση σχετικά, διότι βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης ε, ε, μπορεί να έχει σημασία αυτό όντως και να έχει την επιλογή και ο πιο αδύνατος. Αλλά και συνήθως το πιο αδύνατο μέρος, ε, ο πιο αδύναμος σύζυγος εδώ είναι η γυναίκα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, όχι απλώς επειδή είμαι γυναίκα εγώ, αλλά επειδή βρίσκεται συχνά σε ασθενέστερη θέση. Και... Πάντα, επειδή υπάρχει αυτή η σχέση εξουσίας, έχεις ένα δυνατό και ένα αδύναμο, δεν θα πρέπει να επιβάλλει τη γνώμη του ο ισχυρό που συνήθω είναι ο άντρα. Επειδή θέλει να ξεφορτωθεί εδώ εισαγωγικών των άλλων. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να μην το ξεχνούμε ποτέ. Αλλά και πάλι στο άρθρο 3 γίνεται λόγος για αυτή την ενημέρωση το informed consent, να ξέρουν τι κάνουν και όχι να είναι ο ένας που έχει τις καλύτερες δυνατότητες και προσβάσεις να ενημερώνεται πώς έχει το δίκαιο σε κάποια χώρα και να επιλέγει και ο άλλος που να μην έχει ιδέα να, να είναι σε ασενέστερη θέση. Αυτό θέλω να αποφύγω εγώ. Έτσι. Είμαστε σε καλό δρόμο και ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις που κάνατε και θα τα κοιτάξω, σας είπα και θα σας πω. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Ευχαριστούμε κυρία Γκέμπχαρτ. Λοιπόν, αυτά για αυτό το σημείο. Έμαθα ότι το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα για την έγκριση της νομοδότησης είναι 27 Σεπτεμβρίου και εμείς θα ψηφίσουμε στις 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου. Συμφωνείτε? Ευχαριστούμε. Α, το επόμενο τότε, το επόμενο. Το 11, δηλαδή τροποποίηση του κανονισμού αριθμός 539 κάθετος 2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών Η υπήκοοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή η τελεία. Η συγγήτρια είναι η κυρία Τάνια Φαγιόν. Αφορά λοιπόν την πρόταση κανονισμού για απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων στη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Αλβανία μετά από την παρουσίαση που έγινε τέλη Απριλίου στην Επιτροπή μας για τα αποτελέσματα των τεχνικών αποστολών που έγιναν στις χώρες αυτές και η Κομισιόν έκανε πρόταση κανονισμού στις 27 Μαΐου. Τώρα θα μας μιλήσει η Κομισιόν, ο κύριος Δεμπρόβερ, αντιδιευθυντής ή υποδιευθυντής να μας παρουσιάσει την πρόταση αυτή και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας της επόμενης φάσης, ιδιαίτερα τις πρόσθετες αποστολές που προβλέπονται για το καλοκαίρι. Και μετά θα γίνει η συζήτηση με τα μέλη, ο κύριος Ντεμπρόβερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σε θέση να παραμείνω σύντομος ε, κατά την παρουσίαση των προτάσεων αυτών, διότι όπως είπατε και ο ίδιος, προκύπτουν από την ίδια την έκθεση που είχαμε την ευκαιρία να υποβάλουμε στην Επιτροπή σας και κλεισμένων των θυρών τον περασμένο Απρίλιο. Αποτελέσματα της αποτίμησής μας είναι ότι είναι αυτό το κείμενο που υποβάλαμε στις 27 Μαΐου, η πρόταση που υποβάλλεται σήμερα στην έγκρισή σας και που στοχεύει στη χορήγηση, σήμα στην κατάργηση της υποχρέωσης θεωρήσεων για τους πολίτες της Βοσνίας και της Αλιβανίας με αντάλλαγμα την κατάληξη, το σεβασμό μάλλον ορισμένων υποχρεώσεων που ακόμη δεν έχουν γίνει σεβαστές. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω εδώ ποια είναι η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα. Ήταν η ίδια για όλες τις χώρες των λεγόμενων Δυτικών Βαλκανίων με τις οποίες η Θεσσαλονίκη Ένωση είχε αναλάβει σοβαρές δεσμεύσεις και βασίζεται σε οδικούς χάρτας με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει και όρους που πρέπει να πληρούν οι χώρες που θέλουν να λάβουν μέρος στη διαδικασία αυτή. Συμπέρασμα λοιπόν της αποτίμησής μας είναι, της αξιολόγησής μας, ότι ήρθε η ώρα να καταργηθούν οι θεωρήσεις οι λεγόμενες βίζες, αλλά με μία ενδιάμεση φάση, δηλαδή πρέπει πρώτα να γίνει μια επαλήθευση των προόδων που θα είχαν γίνει επί τριών κριτηρίων. Για την Αλβανία, την ανάπτυξη μιας πολιτικής για τις επιστροφές Αλβανών στην Αλβανία, την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων της εφαρμογής του νομικού πλαισίου καταπολέμησης του οργανωμένου εγκαλήματος και της δωροδοκίας ή διαφθοράς και την πραγματική εφαρμογή, αποτελεσματική εφαρμογή των όσων είχαν αποφασιστεί για τα κατασχέσεις των κερδο, παρανόμων κερδών του οργανωμένου εγκουλήματος και άλλα τρία κριτήρια για τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη. Πρώτον είναι σαν της Αλβανίας δηλαδή την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων εφαρμογής του πλαισίου καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς ιδωροδοκίας και τα δύο υπόλοιπα είναι ειδικά για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, εναρμόνιση της, νομοθεσ... της ε, νομοθεσίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος για τον ΠΡΚΟ με την ισχύουσα νομοθεσία πανομοσπονδιακός και εφαρμογή προοδευτική εφαρμογή βέβαια, του σχέδιου δράσης που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2010 σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αστυνομικών αρχών και υπουργείων. Τα κριτήρια αυτά είναι σαφή, ο, αντικειμενικά και τα συμπεράσματα αυτά τα δέχτηκαν και οι αλβανικές και οι βοσνιακές αρχές. Η επαλήθευση του κατά πόσον ε, υπήρξε πρόοδος θα γίνει. Θα γίνει μέσω της διοργάνωσης αποστολών εμπειρογονωμόνων. Εν καιρό το δέοντι και εν ευθέτω χρόνο όπως θα καθοριστεί από κοινού με τις αρχές των χωρών αυτών. Με στόχο να καταφέρουμε χάρη στις προόδους που θα έχουν γίνει να δείχνουν οι μελέτες αυτές λοιπόν από τις αποστολές ότι τα κριτήρια που είχαμε θέσει έχουν εφαρμοστεί και επιτευχθεί. Προσωρινές ημερομηνίες έχουν ήδη καθοριστεί για τις αποστολές αυτές. 5 με 8 Ιουλίου για την Βοσνία και 8 με 15 για την Αλβανία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι ακόμη προσωρινές και πρέπει να επιβεβαιωθούν από κοινού και με βάση πληροφορίες που δεν έχουμε ακόμα. Πριν το τέλος της εβδομάδας όμως θα τις έχουμε. Αν το χρονοδιάγραμμα αυτό εγκριθεί και εφαρμοστεί, τότε θα είμαστε μάλλον σε θέση να υποβάλουμε στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές Σεπτεμβρίου την αξιολόγησή μας, αξιολόγηση της Κομισιόν, με βάση τις αποστολές αυτές και τα συμπεράσματα των εμπειρογονωμόνων. Και τότε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφανθούν γνωρίζοντας τα πράγματα, πώς έχουν τα πράγματα. Ας επαναλάβω όμως ακόμη μια φορά κύριε Πρόεδρε ότι εδώ πρόκειται για αντικειμενική αυστηρή διαδικασία που στοχεύει στην επίτευξη ενός κύριου πολιτικού στόχου τον οποίο κανείς δεν αμφισβητεί. Δηλαδή την εφαρμογή των πολιτικών δεσμεύσεων που είχαμε αναλάβει για τις χώρες των δυτικών λεγόμενων Βαλκανίων, όπως είχε γίνει για τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Να εφαρμοστεί δηλαδή να δημιουργηθεί ένας χώρος ελεύθερης διακίνησης χωρίς τουλάχιστον την ανάγκη των θεωρήσεων πρέπει να τονίσω ότι καθόλου είναι αυτή τη διαδικασία εμείς ως Κομισιόν ε, απολαύσαμε πλήρη ελευθερία για τις μετακινήσεις μας στις χώρες αυτές και πέρα από τις ε, πολιτικές τους υπηρεσίες, από το σύνολο των κυβερνήσεών τους είχαμε πολύ καλή μεταχείριση. Γενικότερα, δεν έχει ακόμα λήξει βέβαια η διαδικασία, αλλά το μάθημα που παίρνουμε μέχρι τώρα από όλα αυτά είναι ότι, ότι η μέθοδος αυτή αποτέλεσε μοχλό για τον πολλαπλασιασμό των μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές για την ασφάλεια των διαβατηρίων, για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και την καταπολέμηση των σάνησης ε, μεταχείρισης. Σε όλα αυτά έχουν γίνει θεαματικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές με την υποστήριξη βέβαια της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιτευχθεί αυτός ο βασικός στόχος της κατάργησης των θεαρίσεων. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, αν και δεν είμαστε ακόμη στο τέλος του δρόμου αυτού και πρέπει ακόμη να περάσουμε από ορισμένε τελικές φάσεις, δεν αμφιβάλλουμε για την ειλικρίνεια των προθέσεων των χωρών αυτών να επιτύχουν την πρόκληση αυτή, να αντιμετωπίσουν την πρόκληση αυτή και η αυστηρή και αντικειμενική μας μέθοδος μέχρι τώρα θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της διαδικασίας και ελπίζουμε, επαναλαμβάνω, να υποβάλουμε το Σεπτέμβριο στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την τελική μας αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Ντεμπάουερ. Πριν μιλήσουν άλλοι από την Κομισιόν, ίσως η Προεδρία, η Προεδρία, ή μάλλον πριν μιλήσουν οι συνάδελφοι, η πρόσωπος της Προεδρίας η κυρία Ζούστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω, ξέρετε ότι έχουμε δεσμευτεί όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και ε, ως μέλος Συμβουλίου και ως Προεδρία, οπότε ε, σήμερα κιόλα με μεγάλη ικανοποίηση ε, είδαμε ότι από την Σουηδία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συνετάχθησαν σε εκείνο τον κατάλογο των χωρών των οποίων οι χώρες δικαιούνται αυτή την θεώρηση για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε χαιρετίζουμε τις προσπάθειες των αυτών των χωρών, ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος εκείνος και στα πλαίσια αυτά ε, καλωσορίζουμε σήμερα όλες αυτές τις προσπάθειες για τις μεταρρυθμίσεις που εξήγησε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ε, προσπάθεια σε σχέση με Αλβανία και Βοσνία, τόσο ώστε να είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει αυτή την πρόταση 27 Μαΐου για να ε, υπάρχουν θεωρίε διαβατηρίων στι χώρε Σέγγεν και για αυτέ τι δύο χώρε. Και εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι η Αλβανία και η Βοσνία Ερτσεχοβίνη πρόκειται να διεκπαιρεώσουν τη διαδικασία ε, ούτω ώστε να είναι δυνατόν να γίνει η των εγγράφων που χρειάζονται και έτσι Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να αποφασίσουν αυτό το οποίο πρέπει να γίνει ούτω ώστε οι πολίτε των δύο αυτών χωρών να μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτή την κατάρριξη τη θεώρηση διαβατηρίου. Η, η Υπουργή Δικαιοσύνη Ιστορικών στο Λουξεμβούργο συνήλθαν στο Λουξεμβούργο και σήμερα μόλις το πρωί έγινε συζήτηση των εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια και στο περιθώριο του Συμβουλίου και Περιμένουμε πώ και πώ τα αποτελέσματα, την αξιολόγηση τη αποστολή των εμπειρογνωμών επί τόπου στι χώρε εκείνε που για να διαπιστώσουν μέχρι ποιο βαθμό έχουν τηρηθεί τα υπεσχημένα, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τώρα θα ακούσουμε τον εισηγητή, την εισηγήτρια, την κυρία Τάνια Φαγιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα αποφάσισα να μιλήσω σλοβενικά για αλλαγή, έτσι μια που παίζει και η Σλοβενία. Εμείς ε, έχουμε μεγάλα πατριωτικά αισθήματα αυτή τη στιγμή. Τελειώνει το μάτς κατά της Αγγλίας και χάνουμε κιόλα και ξυπνάει έτσι το σλοβενικό μέσα μας. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω στα σλοβενικά και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για τις παρουσιάσεις τους. Ήταν εκτενέστατες και είμαι εισηγήτρια για τη Βοσνία, Ζεγοβίνη και την Αλβανία και χαίρομαι ιδιαίτερως ε, που βλέπω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέτει νομοθετική πρόταση την κατέθεσε τέλη Μαΐου για την ε, κατάργηση των θεωρήσεων διαβατηρίου. Δεν μπορώ παρά να σας ευχαριστήσω ε, για την τόσο καλή συνεργασία με την Κομισιόν, την Ισπανική Προεδρία και τους κοιόδης συγητές. Επίσης θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους ιδιαιτέρως τις αρχές της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης καθώς και της Αλβανίας. Για τη δική μας Επιτροπή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι η διαδικασία απελευθέρωσης των θεωρήσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και εδώ συμπεριλαμβάνω και το κράτος του Κόσοβου που ε, είναι προς το παρόν εκτός του διαλόγου για τις θεωρήσεις. Είναι στα τελικά στάδια και η Βοσνία, η Ζεγοπίνη και η Αλβανία. Και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το παραδέχθηκε. Ότι και τα δύο κράτη έχουν ε, καταβάλει σημαντικά βήματα προόδου ε, τους τελευταίους μήνες και Ελπίζω οι ειδικοί εμπειρογνώμονε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισκεφθούν πριν από το καλοκαίρι και τι δύο χώρε για να τα διαπιστώσουν δύο όμαση. Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι και οι δύο χώρε είναι έτοιμε και οι δύο δηλώνουν ότι πληρούν όλα τα κριτήρια. Συμφωνώ βέβαια ότι ε, αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις και θα πρέπει βεβαίως να το απληρούν και οι δύο χώρες για να απελευθερωθεί η διαδικασία αυτή θεώρησης των διαβατηρίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το βήμα αυτό, ιδιαίτερα για νέους της περιοχής που θέλουν να ταξιδεύουν, διότι οι νέοι περιμένουν να έχουν την ευκαιρία να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμιά φορά φοβούμε ότι ξεχνούμε το γεγονός ότι οι χώρες αυτές είναι στην άμεση γειτονία μας και περιμένουν διακαώς να έχουν την ευκαιρία να ταξιδεύουν οι πολίτες, να έρθουν πιο κοντά στην Ευρώπη. Ζούμε καιρούς ε, οικονομικής κρίσης και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην θέλει ε, πια άλλες διευρύνσεις. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση και πολιτικό στένος και θάρρος για να ανοίξουμε τις θύρες μας προς τους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων. Ιδιαίτερα τη στιγμή που πληρούν, όπως είπαμε, όλα τα απαραίτητα κριτήρια. Έχω όμως και μία ερώτηση. Να σας πω. Όταν καταθέσαμε την πρόταση αυτή, γιατί δεν βάλαμε και καμιά ημερομηνία. Πέρυσι τον Ιούλιο η Σερβία, το Μαυροβούνιο και δεν θυμάμαι ποιος άλλος, μια άλλη χώρα ακόμα, έλαβαν ημερομηνία για την 1η Ιανουαρίου του 2010. Τώρα, αυτή τη φορά δεν έχουμε βάλει. Για ποιο λόγο δεν το κάναμε αυτό για τη Βοσνία και την Αλβανία, μπορείτε να μου εξηγήσετε σας παρακαλώ. Υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν αντιλαμβάνομαι. Mm. Ας βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα και για τις χώρες αυτές χρειάζονται κίνητρα και χρονικά. Είμαστε πλέον στα τεχνικά στάδια της διαδικασίας. Αλλά εκτός από τεχνικό είναι και πολιτικό το θέμα. Και ε, ξέρετε ότι είναι μεγάλη ένταση, ιδιαίτερα στη Βοσνία Ζεγοβίνη, όπου το φθινόπωρο επίκυνται εκλογέ. Και όλη η πολιτική ε, προεκλογική εκστρατεία είναι στο Ζενίθ. Τελικά, όμως, αν δεν έχουμε αποτελέσματα θα πληγεί ο λαός. Στην Αλβανία επίσης είναι πάρα πολύ τεταμένα τα πράγματα. Και ακριβώς επειδή υπάρχει τόση ένταση, ίσως θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει. Είπαμε ότι η Ένωση υποφέρει από την κόπωση της διεύρυνσης, αλλά δεν θέλω να κλείσουμε τις πόρτες των θεωρήσεων προς τα Δυτικά Βαλκάνια, ούτε να υψώσουμε νέα τύχη προς τους λαούς αυτούς. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην παρούσα Επιτροπή να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ψηφίσουμε την έκθεση το Σεπτέμβριο. Αν γίνεται αμέσως μετά την δημοσίευση της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων για την πρόοδο. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν είναι δυνατόν, να έχει την αξιολόγηση ε, και να μας τη φέρει στις 3 Σεπτεμβρίου που θα συνεδριάσουμε για πρώτη φορά για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στη δεύτερη ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Αν το κάνουμε αυτό, ε, διατηρούμε την προσήλωσή μας και τη δεσμευσή μας προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους δώσουμε προτεραιότητα θα πρέπει να μην αθετήσουμε το λόγο μας. Έχουμε δώσει το λόγο μας, θα πρέπει να τον τηρήσουμε. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να έρθουν εδώ να ζητήσουν άσυλο, να πάρουν τις δουλειές μας. Θα πρέπει να γκρεμίσουμε τα τείχη των θεωρήσεων για να μπορεί ε, ο κόσμος να ταξιδεύει ελεύθερα και οι νέοι να γνωρίσουν και να καταλάβουν τις ευρωπαϊκές αξίες για να μην απομακρυνθούν και στρίψουν την πλάτη τους στην Ευρώπη. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια το σύντομότερο. Ευχαριστώ. Thank you. Now, Mrs. Uh, Ευχαριστώ κυρία Κοράτσα Μπίλτ, σκιώδης. Also... Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να χαιρετήσω την πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την ε, ε, Βοσνία και την Αλβανία το να μπορούν να μπουν στην ε, ζώνη Σέγγεν. Θα πρέπει βεβαίω επίση να περάσουμε τι χώρε εκείνε για την πρόοδο που πέτυχαν. είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο πέτυχαν και για αυτού και για την ευρωπαϊκή του προοπτική. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο αυτή η βίζα, είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες για την κοινωνία αυτή, για το μέλλον τους σαν, για το, για, για, το μέλλον τους σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Οπότε δεν θα πρέπει και εμείς παρά ε, θα πρέπει να, να βεβαιώσουμε το ότι δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία που θα γίνει στο Κοινοβούλιο και με μεγάλη μου χαρά σας λέω ότι συνοήθηκα με την εισηγήτρια, συμφωνώ με το χρονοδιάγραμμα που αυτή όρισε και περιμένουμε την ε, έκθεση πεπραγμένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να, να δουν όλα αυτά τα πραγματικά περιστατικά που γίνουν, τα στοιχεία, να, να δούμε αν τα κριτήρια πληρούνται και θα έπρεπε να τα ίδια κριτήρια αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί τις άλλες τρεις χώρες. Και ακολούθησαν αυτή τη διαδικασία τις άλλες χώρες και τα συμφωνήσαμε πρωτού, πριν, πριν ολοκληρωθεί η διαδρομή. Επομένω. θέλουμε να ξέρουν οι λαοί αυτοί ότι θέλουμε να φτάσουμε στο τέλο τη διαδρομή. Πρόεδρε, θα συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία μας με την Κομισιόν, την εισηγήτρια, του άλλου συναδέλφους, τόσο ώστε το πολύ μέχρι το τέλο τη χρονιά να έχουμε πετύχει η Γερμανία και η Βοσνία την κατάρριξη της ε, βίζα. Από... Για να δούμε. Ποιος η κυρία Ρασαρτζεντίνη, όχι. Όχι, η κυρία Μποσκιούρτ. Μποσκιούρτ, yes. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας πω και εγώ σύντομα την άποψή μου. Όπως και η συγκήτρια, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Έχω πάει και εγώ στην Βοσνία πριν από καιρό. Πράγματι η νεολαία θέλει να βγει από την απομόνωσή της. Και θα ήταν καλό να μπορούν να ταξιδεύουν εύκολα. Και πέρυσι ήδη σε ένα ψήφισμα ζητούσαμε από την Κομισιόν να βοηθήσει τη Βοσνία όσο το δυνατόν συντομότερα για να ετοιμαστεί για την προενταξιακή της διαδικασία. Και συμφωνώ και με την κυρία Κοράτσα Μπίλτ που λέει ότι πρέπει να εφαρμοστούν τα ίδια κριτήρια όπως και για τις άλλες τρεις χώρες ως προς τον καθορισμό ημερομηνία. Πρέπει να δώσουμε ημερομηνία στη Βοσνία. Ελπίζω στη δεύτερη σύνοδο του Σεπτεμβρίου να μπορέσουμε να ψηφίσουμε από αυτό. Αυτό θα, έδινε, θα ήταν μια πολύ καλή χειρονομία έτσι ώστε να δώσουμε επιτέλους μια ευρωπαϊκή προοπτική στη Βοσνία. Μόνο έτσι οι χώρες αυτές των Βαλκανίων θα μπορέσουν να ανοικοδομηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπουζουτήλ. Ευχαριστώ πρόεδρε, συντομότατα. Υποστηρίζω όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, ιδιαίτερα ως προς τον καθορισμό ημερομηνία. Αλλά θέλω επίση να τονίσω την ιστορική σημασία που έχει αυτή η συνεδρίαση όπου λείπουν τόσοι βουλευτές. Για μας η Βοσνία μπορεί να φαίνεται ασήμαντη γιατί θεωρούμε σαν δεδομένη την ελεύθερη διακίνηση επειδή την έχουμε αλλά για τους πολίτες της Αλβανίας και της Βοσνίας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και η απελευθέρωση των θεωρήσεων θα ήταν όντως το πρώτο βήμα για την ευρωπαϊκή τους ολοκλήρωση. Πρέπει όμως και εμείς να καταλάβουμε τη σημασία που έχει αυτή η συζητησούλα μας εδώ για εκείνους. Ίσως πολλοί από αυτούς να παρακολουθούν τη συζήτηση με τεράστιο ενδιαφέρον διότι θα έχει διαφορά στη ζωή τους. Θα αλλάξει η ζωή τους από αυτά που θα αποφασίσουμε. Και καταλήγω με μία έκκληση για φρόνηση ιδιαίτερα στις αρχές των χωρών αυτών. Δεν σημαίνουν όλα αυτά ότι η ελεύθερη διακίνηση θα εφαρμοστεί όπως εμείς μέσα στην Ένωση και δεν πρέπει να τους το λέμε γιατί τους παραπλανούμε. Δεν σημαίνει ότι μπορούν να πηγαίνουν ελεύθερα όντως στην Ευρώπη να κατοικήσουν και να σπουδάσουν. Ελπίζουμε κάποτε να φτάσουν και εκεί αλλά δεν είναι αυτό το βήμα που συζητάμε σήμερα. Και άρα είναι σημαντικό να μην δημιουργήσουμε φρούδες ελπίδες αλλά να τους εξηγήσουμε τι ακριβ, περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Ευχαριστούμε κύριε Μπουζουτήλ. Η Επιτροπή μας είτε με λίγους είτε με πολλούς κάνει πάντα τη δουλειά της η οποία έχει τη σημασία που γνωρίζετε. Έχουν ασκηθεί ερωτήματα προς την Κομισιόν, ας απαντήσει ο κύριος Δεμπράουερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την άδειά σας θα απαντήσω σε τρία ερωτήματα. Πρώτον η Κομισιόν πράγματι δεν έχει ακόμη καθορίσει την τελική ημερομηνία για την κατάργηση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Δεν είναι γιατί το ξεχάσαμε. Mm. Εσκεμένα το κάναμε. Γιατί η κατάργηση του καθεστώτος των θεωρήσεων θα γίνει όταν θα έχουν πληρωθεί τα τρία κριτήρια που ανέφερα. Και όταν ο νομοθέτης, δηλαδή εσείς και το Συμβούλιο, θα θεωρήσει ότι με βάση την αξιολόγησή μας πράγματι επληρώθησαν τα κριτήρια. Στα χέρια λοιπόν του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εναπόκειται όταν θα έχει λάβει την αξιολόγησή μας να αποφασίσει το πότε θα εφαρμοστεί η κατάργηση των θεωρήσεων ακριβώς. Δεύτερον, για την αξιολόγηση την έκθεσή μας. Η κυρία Φοκέ μας είπε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου μπορεί να τη συζητήσετε. Εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας υποσχεθώ εξ ονόματος της Κομισιόν ότι θα έχετε έκθεση γραμμένη μέχρι τότε. Νομίζω όμως ότι αν θέλει και η δική σας επιτροπή θα μπορούσαμε στις 3 Σεπτεμβρίου, την 3η Σεπτεμβρίου δηλαδή, προφορικά να σας αναφέρουμε τα κύρια συμπεράσματα της αξιολόγησής μας. Της οποία η γραπτή μορφή θα σας υποβληθεί αργότερα. Τρίτον κύριε Πρόεδρε και πολύ σημαντικό. Όπως είπαν και πολλοί άλλοι, ιδιαίτερα δε ο κύριος Μουσουτήλ, ποια είναι ακριβώς η σημασία της κατάργησης του καθεστώτος των θεαρήσεων Σέγγεν βραχέας διαρκείας. Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Βραχίας, βραχίας, όχι βραχίας. Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών, Αλβανία, Βοσνία, γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι η σημασία αυτή ακριβώς, είναι όπως είπε ο κύριος Μουζουτήλ, δηλαδή οι αρχές των χωρών αυτών έκαναν καμπάνιες πληροφόρησης για να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις αναφέροντας συγκεκριμένα ποια δικαιώματα θα έχουν θα απορρέουν από την κατάργηση του καθεστώτος αυτού, αλλά και ποια όρια έχουν τα δικαιώματα αυτά, τι θα είναι δυνατόν και τι δεν θα είναι δυνατόν μετά την κατάργηση. Αυτό είναι ουσιοδέστατο και για μας είναι πολύ σημαντικές οι καμπάνιες αυτές που έκαναν οι δύο κυβερνήσεις. Γιατί στις αρχές του χρόνου είχαν αρχίσει παρεξηγήσεις οι οποίες μετά λύθηκαν βέβαια από τις ίδιες τις κυβερνήσεις δεν είχε καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι σήμαινε η κατάργηση της βίζας Στέγγεν. Αλλά με τις καμπάνιες αυτές και, από την και στην Αλβανία και στη Βοσνία ησυχάσαμε. Και θεωρούμε τώρα ότι οι παρεξηγήσεις που για σύντομο χρονικό διάστημα είχαμε γνωρίσει στις αρχές του χρόνου δεν θα επαναληφθούν. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστούμε και πάλι κύριε Ντεμπράουερ. Κανένα άλλο σχόλιο ή καμιά αντίδραση. Μήπως η κυρία ειπε η Ευχαριστώ πολύ για τις επιπλέον διευκρινήσεις σας και εγώ. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι αν είναι δυνατόν μετά την ολοκλήρωση του έργου των αρχίσει αρχές βρίου. θέλουμε, εάν είναι δυνατόν, ε, να καθορίσει τα πολιτικά του, συνεχίζουμε και θέλουμε το κείμενο. Πάρα πολύ σωστά αυτό που είπατε για την ημερολογική εκστρατεία και στις δύο χώρες. Προσπαθούμε να συνειδητοποιήσει ο κόσμος όσο γίνεται περισσότερο το τι γίνεται, να ξέρει ο κόσμος ότι πρόκειται για ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων με κάποιες κάποιους περιορισμούς. Όλοι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το χρονοδιάγραμμα, κυρίως τι πρέπει να γίνει πριν τις θερινές διακοπές, γιατί πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε καθορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Τώρα δεν έχουμε, οπότε δεν έχω καταλάβει. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Επομένω, από τη... πάμε στη... τον Ιούλιο, θα υπάρχει σχέδιο κειμένο από την εισηγήτρια 12 και 13 Ιουλίου συγκεκριμένο οπότε θα έχουμε τον καθορισμό της ε, προθεσμίας για την έκθεση, διότι η διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί μετά τις στενές διακοπές, οπότε πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι το υπαριθμό 12. Το 12 αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολισμού 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Τμήμα 3. Επιτροπή. Διάρεμη. Και έχουμε τώρα το δεύτερο έγγραφο εργασία για τον προπολισμό για τη χρήση 2011. Πρώτη έγγραφο το οποίο προφανώ μα έχει συντάξει ω πρώτης επιτροπή. Νομίζω έχετε λάβει το σχέδιο κειμένου και θα προσπαθήσω να σας πω σε αδρές γραμμές τα βασικά στοιχεία αυτής της γνωμοδότησης Como Πρόκειται για το σχέδιο κειμένου αυτή τη γνωμοδότηση. που πρέπει να διεκπεριώσουμε και αφορά την Επιτροπή μα. Και να απευθύνομαι δε αυτή μας την έκθεση στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών και έχουμε εδώ ε, προσεκτημένες τις ε, τροπολογίες που αφορούν τον προϋπολογισμό. Discutir en la próxima reunión libre del 12 y 13 de Όλα αυτά θα συζητηθούν 12 και 13 Ιουλίου που είναι η επόμενη συνάντησή μα. Η ψηφοφορία θα γίνει στι 2 Σεπτεμβρίου. Γιατί η μοναδική δυνατότητα που μα παρέχεται είναι αυτή. Ξέρετε, θα πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή των Προπολογισμών αυτή η έκθεση στι 8 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε μόνο μία συνάντηση πριν τι 8 και 9. Έχουμε συνάντηση 12 Σεπτεμβρίου. Οπότε θα πρέπει να μεταφραστούν όλες οι τροπολογίες και όλες τις επίσημες γλώσσες για να γίνει η ψηφοφορία. 18 de Άρα θα πρέπει να έχουμε κάνει δουλειά μα πριν έρθει η ώρα των διακοπών και εάν πάντω συμφωνείτε να μην έχουμε όλε τι μεταφράσει θα μπορούσαμε να πάει 26 Αυγούστου η προθεσμία για τι ε, τροπολογίε. 26 Αυγούστου το μεσημέρι. Ούτω ώστε να μπορέσουμε ε, να έχουμε ε, τελειώσει πριν να ξαναρχίσει το, η συνήθις ε, πορεία του κοινοβουλευτικού έργου. Οπότε. Αυτό θα πούμε. Η προθεσμία είναι 26 Αυγούστου το μεσημέρι, αφού δεν υπάρχει κάποια ένσταση. Επί του ουσίας τώρα... Έχετε το συνοδευτικό κείμενο, το επεξηγηματικό. Ξέρετε πώς έχουν τα πράγματα. Κινούμεθα σε ένα πλαίσιο χρηματοπιστωτικής κρίσης. Είναι κάτι που έχει χτυπήσει όλα τα κρατημέλια. Οπότε Γι' αυτό και μιλούμε για κάποιους είδου περικοπές στον προπολογισμό. Το Συμβούλιο πρώτον προβεί σε περικοπές για τη χρήση 2011. Άρα και εμείς θα πρέπει με μεγάλη επιφύλαξη να δούμε ποιες είναι οι δικές μας προτεραιότητες. Όπως γνωρίζετε έχουμε κάποιες προσευχές δράσεις και προγράμματα πιλωτικά για τα οποία έχουμε λάβει 14 προτάσει. Περισσότερο από την περσινή χρήση. Πέρσι είχαμε μόνο δύο προπροσκευαστικές δράσεις και μόνο ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Όσον αφορά τι δικέ μα ομοδιότητες. Επομένως, τώρα θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητες, διότι δεν είναι δυνατόν να εγκριθούν όλες αυτές οι δράσεις, οι προπροσκευαστικές και όλα τα προγράμματα. Όσον αφορά τώρα τα προγράμματα νομίζω ότι αξίζει εδώ να κάνουμε μια ειδική μνήμα εις τρεις διατάξεις. Πρώτον, ω συνήθως όσον αφορά την Frontex. Ε, θα γίνει αναθεώρηση του κανονισμού για αγορά υλικού. χτενιστεί Επομένως το κεφάλαιο μας αφορά, αλλά ε, ζητούν να υπάρχει ένα ποσό αποθεματικού το οποίο να εκταμιεύεται εάν το ζητήσει η υπηρεσία, η Frontex. Σε και θέσει που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού. Εάν υπάρχει πρόβλημα απορρόφησης ή εκταμίευσης των προβλεπωμένων κονδυλίων. Έχουν ζητήσει αύξηση σημαντική. Δεν νομίζω ότι θα είναι δυνατόν να μπορούμε να καλύψουμε αυτό το αίτημα, γιατί είναι μεγάλο ποσό. Αλλά αξίζει να προσπαθήσουμε κάτι να κάνουμε όσον αφορά την υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί βρίσκεται σε φάση πάρα πολύ σημαντική τη ζωή τη. Μιλάμε για ένα 50% αύξηση. 5%, 5%, αύξηση. Και επομένως να κάνουμε εδώ κάποιες τροπολογίες, ούτω ώστε να γίνει αυτή η αύξηση του προπολογισμού. Επομένως, είμαστε ανοιχτοί στο αίτημα αυτό Επομένω, θέλω να λάβουμε υπόψη αυτό το αίτημα. Τώρα, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Ο πρόεδρο τη ομάδα του άρθρου 29, όπω και ο προηγούμενο πρόεδρο, ο προκάτοχό του, ζητούν και οι δύο να λάβουμε υπόψη την δύσκολη οικονομική κατάσταση όσον αφορά την ομάδα για το άρθρο 29 για να επιτελέσουν το έργο τους και ζητούν τη βοήθειά μας. Εάν συμφωνούν οι συνάδελφοι, θα πρέπει και εδώ να γίνει μια αύξηση της πρικοδότησης όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Επομένως θα πρέπει να ζητηθεί μια λύση σε συνεργασία με τις αρμοδίες υπηρεσίες. Να δούμε τι προτάσεις έχουμε τι προτάσεις ε, έχετε να μου πείτε, γιατί τώρα θα κάνουμε ένα γύρο τραπέζι και μπορείτε να λάβετε το λόγο. Για να συζητήσουμε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης, γιατί θα πρέπει κάπου να καταλήξουμε να ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Παγιέτ είναι εδώ, ναι, σηκώνει το χέρι της. Παρακαλώ, Πέστε μα την άποψη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας αυτή και την παρουσίαση. Μερικά εισαγωγικά σημεία, αν μου επιτρέπετε. Σε ό,τι αφορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά ε, προγράμματα, δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω το υπογραμμίσω λέω την υποστήριξή μας. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι στο πλαίσιο των υφισταμένων προγραμμάτων έχουμε είτε δυνατότητα κοινοτικής δράσης είτε τεχνικής ε, οικονομικής βοήθειας έτσι ώστε να χρηματοδοτούμε σε ορισμένες περιπτώσεις μερικές από τις δράσεις αυτές. Ενώ άλλα προγράμματα προβλέπουν ήδη τέτοιες δράσεις ε, που ανταποκρίνονται στι επιθυμίες σας για τις προπαρασκευαστικές δράσεις στα πιλωτικά προγράμματα. Είδαμε τις προτάσεις σας. Θα τα υποβάλουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες και για τον προϋπολογισμό. Και πάλι θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποια είναι η προστιθέμενη αξία, η υπεραξία στα ήδη υφιστάμενα προγράμματα και να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες του προπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τη Frontex, αν θέλετε να σας δώσω κάποια εξήγηση για το πώς έγινε το αίτημά μας ως προς το δημοσιονομικό σκέλος. Όπως γνωρίζετε, λαμβάνουμε υπόψη πώς να το πω αυτό. Ε, λαμβάνουμε υπόψη τις δημοσιονομικές προοπτικές και το συνολικό ποσό που προβλέπεται με ένα συγκεκριμένο περιθώριο και μια συγκεκριμένη οροφή. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ε, στους υπολογισμούς που κάνουμε για τις πιστώσεις και τα σχετικά αιτήματα λαμβάνουμε υπόψη τι δεν έχει δαπανηθεί, τι δεν έχει απορροφηθεί στην προηγούμενη χρήση. Δηλαδή, στις πιστώσεις πληρωμών συγκεκριμένα, ακριβώς θα πρέπει να προσθέτουμε αυτά τα ποσά ε, που προστίθεται στις πιστώσεις στις φετινές. Δηλαδή ότι πλεόνασμα έχουμε από το προηγούμενο οικονομικό έτος. Έτσι υπολογίζεται ο προεπλογισμός. 85 και εκατομμύρια ήταν για το 2010 και ζητούμε 80 για το 2011. Θυμίζω ότι η αρχική μας ε, πρόταση ήταν 80,55 και είχε προσθέσει η Δημοσιονομική Αρχή πέρυσι 5 εκατομμύρια επιπλέον. Και τώρα έχουμε βεβαίως ε, πλεόνασμα περίπου 6 εκατομμύριων ευρώ με αποθέματα που θα πρέπει να απορροφηθούν πριν ε, αντλήσουμε άλλες πιστώσεις πληρωμών. Επίσης ζητήσαμε πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων, ε, του οργανογράμματος μάλλον, γιατί δεν έχουν πληρωθεί οι θέσεις στο Frontex. 44 θέσεις χειρεύουν. Λοιπόν, επειδή χειρεύουν αυτές οι θέσεις, παγώνει το, το οργανόγραμμα, συγγνώμη, ε, να δούμε όμως ε, τι θα γίνει με τις λειτουργικέ ε, δαπάνες που αυξάνονται και εν ώψη της πρώτας αναθεώρησης του Frontex που συζητείται αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, να βάλουμε στο αποθεματικό ένα ποσό, νομίζω είναι η σωστή προσέγγιση αυτή, για να μπορέσουμε ταυτόχρονα να δούμε πώ απορροφώνται τα κονδύλια, πώς ε, εξελίσσονται τα πράγματα και να δούμε εν ευθέτω χρόνο αν όλα αυτά μπορούν να ξαναμπούν στο κονδύλι στη θέση του προπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, συμφωνώ με τη συνετή σας προσέγγιση, τη συμμερίζομαι και εγώ, όπως και με το Frontex, ακολουθούμε τα ποσά που προβλέπονται από τις δημοσιονομικές προοπτικές. Από την άλλη βέβαια είναι επίσης γεγονός ότι ο οργανισμός αυτός θα απορροφήσει καλά τα κονδύλια του, καλό είναι και αυτό, και δεν μπορούμε παρά να είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι και να συμφωνούμε με τις εργασίες που κάνει ο οργανισμός αυτός ως προς τη συλλογή δεδομένων και στοιχείων. Σε γενικές γραμμές λοιπόν δεν έχουμε ούτε επιφυλάξεις ούτε αντιρρήσεις για την αύξηση της χρηματοδότησης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο βαθμό που ε, μένουν, παραμένουν σε ένα λογικό πλαίσιο και απαντούν σε πραγματικές ανάγκες που έχει καταδείξει ο οργανισμός αυτός. Επίσης, από πλευρά μας, Εξετάζουμε τη δυνατότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης καθώς ενσωματώνονται οι δραστηριότητες του τρίτου πυλώνα και οι εκτιμήσεις είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε νομίζω ότι η συνετή και φρόνιμη προσέγγιση σας είναι η ορθή σε ό,τι αφορά την αύξηση των κονδυλίων για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σας υποστηρίζουμε σε αυτή την οδό. Σε ό,τι αφορά τώρα το άρθρο 29 και την αντίστοιχη ομάδα εργασίας, Κατανοώ ότι έχουν ανάγκες και εκείνοι και εμείς είμαστε σε επαφή μαζί τους όπως και εσείς για τη γραμματεία τους προκειμένο. Ωστόσο, πρέπει να θυμίσω ότι μέγα τμήμα της χρηματοδότησης των εργασιών αυτών προέρχεται από το συνολικό προϋπολογισμό που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις γενικές διευθύνσεις, για τα έξοδα εκτός ε, έδρας, συνεδριάσεις, ε, ομάδες εμπειρογνωμόνων και εκεί είναι πάρα πολύ περιορισμένα τα κονδύλια που διαθέτουμε. Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και φρόνιμοι στην, ε, στη διαχείριση γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Ο κύριος Ευχαριστώ στα ισπανικά. Και συνεχίζει Ολλανδικά ο Ε, καταρχάς θα ήθελα να σας απευθύνω τι ευχαριστίες μου καθώς και τα συγχαρητήριά μου για την ισόρροπη έκθεση που συντάξατε. Ε, με τρόπο πάρα πολύ νυφάλαιο και ήρεμο και μετά από μεγάλο προβληματισμό και όρημη σκέψη ε, περιγράφεται πολύ σωστά τον προπολογισμό. Αυτό πρώτο. Έχω μερικές ερωτήσεις τώρα για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Έχω καταλάβει ότι είναι πάρα πολλά τα αιτήματα ε, για να μπουν στα πιλωτικά προγράμματα. Και ρωτώ, ποια στρατηγική έχετε εσείς στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, πώς θα καταφέρετε ε, να ανταποκριθείτε σε νέα αιτήματα. Σε... Πώς θα εγκριθεί μια αίτηση, ας πούμε, να μπει κανείς σε ένα πολιτικό επίλωτικο πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι θα μείνετε με σταυρωμένα τα χέρια. Ε, δεύτερο, οικονομίες. Είπατε εισαγωγικά ότι ενδεχομένω χρειάζονται ε, περικοπές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον προϋπολογισμό για οικονομίες. Μα έχουμε και δυνατότητα συζήτησης για ε, τις προτεραιότητες. Ε, δεν ε, μ' αρέσει ο τρόπος που ακολουθούν στην Ολλανδία που κόβουν την πίτα, που τη μειώνουν την πίτα. Θα πρέπει να έχουμε προτεραιότητες ε, και από εκεί να περικόπτουμε. Και με το Frontex πραγματικά πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Θα πρέπει να ε, εξαντλούν το υπροπολογισμό τους με σωστό τρόπο. Και ένα τελευταίο για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κατανοώ την επιφυλακτικότητά σας, αλλά για μας το 5% είναι ένα πρώτο βήμα. Αν υπάρχουν και άλλες ε, δυνατότητες αύξησης του προϋπολογισμού, θα το υποστηρίξουμε ως ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτά σε πρώτη φάση ως μια πρώτη αντίδραση στη έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Έχω μερικές ε, ερωτήσεις και μερικά σχόλια για ε, τα έγγραφα εργασία σας. Για το πρώτο, στη σελίδα 2 αναφέρετε τις αναλήψεις υποχρεώσεων και στο 8 και μιλάτε για κατεπήγοντα μέτρα για μαζική συρροή ε, προσφύγων, 3,7 εκατομμύρια έχετε βάλει εκεί. Αυτό το ταμείο, εξ όσων γνωρίζω, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε από την ίδρυσή του και μετά, γιατί θεωρείται ακόμα σκόπιμο να υπάρχει και να χρηματοδοτείται. Και για το Frontex, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, Δέκα εκατομμύρια ευρώ δεν έχει απορροφήσει πέρσι ο Frontex. Γιατί? δεν ήταν σε θέση να το απορροφήσουν. Ή μήπω χρειάζονται λιγότερα. Μήπω χρειάζεται περικοπή εκεί αντί για αύξηση. Από ό,τι φαίνεται δεν χρειάζονται επιπλέον χρηματοδότηση αφού δεν τα απορροφούν. Τότε γιατί να του τα δώσουμε. Είναι λογικό, δεν σα φαίνεται. Και στη σελίδα 5, τελευταία σελίδα του έγγραφου εργασία, δεν έχω καταλάβει ακριβώ, τι λέτε εκεί. Επιπλέον 3 εκατομμύρια θα πρέπει να δοθούν στη Frontex από τα έσοδα, revenues λέει εδώ, τι σημαίνει αυτό, αυτό τι εννοείται, ε, το πλεόνασμα του περασμένου έτους ή κάποια άλλα κονδύλια. Και για το δεύτερο έγγραφο εργασίας, α, για τον Οργανισμό θεμελιδών Δικαιωμάτων. Λέτε ότι σας ζητούν περισσότερα χρήματα και βάλατε 5% περισσότερο. Εντάξει, ε, θεωρήσατε σκόπιμο κάτι τέτοιο, αλλά από πού το βγάλατε αυτό, έχετε κάνει εκτίμηση, τι χρειάζεται για τον οργανισμό αυτό μετά τη Λισαβόνα. Γιατί επιλέγετε αυτό το 5% ε. ως σύσταση. Έχουν 5% περισσότερο φόρτο εργασίας. Πού το βρήκατε, από πού το βγάζετε αυτό το 5%. Από πού προκύπτει. Και μπορούμε να έχουμε και με έναν υπολογισμό καλύτερο. Και ένα τελευταίο. Α, ναι. DLS IT και το αντίστοιχο οργανισμό που τα διαχειρίζεται αυτά. Γιατί τόσα πολλά λεφτά, συμφωνώ, για έναν οργανισμό που ακόμα δεν έχει συσταθεί. Περισσότερα από παίρνει το Γραφείο υποστήριξη Προσφύγων που ψηφίσαμε όλοι και καλά κάναμε και το ψηφίσαμε. Αυτός ο οργανισμός ε, για τις τεχνολογίες πληροφορικής ακόμα δεν έχει καν ιδρυθεί για τα δίκτυα. Δηλαδή ούτε λόγο έχουμε επ' αυτού ούτε τίποτα. Γιατί δεν του δώσουμε τόσα χρήματα. Τα μισά είχε πάρει την πρώτη χρονιά λειτουργία στο γραφείο για τους πρόσφυγες. Αυτά. Ο κύριος Μπουσούτιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να προσθέσω μερικά σχόλια ε, επιπλέον των όσων είπε ο συνάδελφός μου Κάμπ προηγουμένως για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Κοιτάζω το έγγραφό σας και βλέπω ότι το 2001 είχαμε τρεις δράσεις και δύο πιλωτικά προγράμματα και το 2010 δύο προπαρασκευαστικές δράσεις και ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Προσοχή! να διατηρήσουμε την παρουσία της Επιτροπής μας ΛΥΜΠΕ σε αυτά τα σημαντικά θέματα και για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται συντονισμός και αυτό ίσως είναι ένα μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε σε όλες τις πολιτικές ομάδες χρειάζεται λίγο συντονισμός για να συμφωνήσουμε και να βεβαιωθούμε ότι παραμένει η παρουσία της ΛΥΜΠΕ της Επιτροπής Εσωτερικών αν δεν συμφωνείτε θα μας αγνοήσει απλούστατα η Επιτροπή ε, Καλό είναι να ακούσουμε τι έχει να πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θα υπάρξουν και άλλα αιτήματα ε, εν ευθέτω χρόνο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσουμε εκεί την συμμετοχή μας και να υπάρχει κοινή δράση και προσέγγιση. Για το Frontex τώρα δεν είμαι βεβαίως ότι συμφωνώ απολύτως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εξής απλούστατο λόγο. Έχουμε αναθεώρηση ε, του κανονισμού για τον οργανισμό και είμαι εγώ εισηγητής και είναι σαφές ότι ο Frontex τώρα επιτέλους ε, θα έχει ιδίους πόρους. Ε, ε, μάλλον θα έχει στοιχεία ενεργητικού τα οποία είτε θα αγοράσει είτε θα νοικιάσει. Ε, και δεν ξέρω, κάπως θα πρέπει αυτό να το ρυθμίσουμε στον επόμενο προπολογισμό, παρά να περιμένουμε να τεθεί σε ισχύ νομοθεσία και μετά να χάσουμε ένα χρόνο και στο 2011 να μην έχουμε χρηματοδότηση. Γιατί δεν θα έχουμε προβλέψει κανένα κονδύλι γι' αυτό. Έτσι, είναι σημαντικό νομίζω και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη Frontex να μας πούν ακριβώς πώς το βλέπουν οικονομικά, πώς το φαντάζονται. Εάν θα πάρουν σάρκα και ως τα αυτές οι θνήσεις που δεν ξέρω είναι ε, πιθανές. Για το γραφείο και πάλι για το άσυλο και τους πρόσφυγες. Από ό,τι ξέρω εγώ δεν έχει διοριστεί καν διευθυντής. Μήπως θα μπορούσε να μας πει περισσότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ε, ψηφίστηκε φέτος προϋπολογισμός και ποιο θα είναι κάπου το χρονοδιάγραμμα, θα έχετε σκεφτεί, για να βεβαιωθούμε ότι θα είναι σε λειτουργία το γραφείο αυτό σίγουρα πριν τα τέλη του έτους. Γιατί δεν έχει νόημα να συζητάμε για τον προϋπολογισμό για το γραφείο αυτό, αν δεν έχει στελεχωθεί και δεν έχει στηθεί και αρχίσει να λειτουργεί. Για τα προγράμματα τα ίδια, για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην αλληλεγγύη, έχουμε ενδιαφέρουσες αυξήσεις ε, για τα σύνορα, για την σωμάτωση, για το Ταμείο Προσφύγων, για την επαναπρόθεση, αλλά ανησυχώ λίγο, ανησυχώ λίγο λέω, γιατί δεν υπάρχει ανάλυση και ε, έλεγχος και αναθεώρηση αυτών των προγραμμάτων, ακόμα και ενημέρωση δεν δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πού πάνε τα χρήματα αυτά που ψηφίζουμε χρόνο με το χρόνο και σε αυτά τα προγράμματα. Πώς χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά, άραγε αρκετά, ε, έχουμε υπεραξία είναι σκόπιμο. Θα θέλαμε πάρα πολύ να τα μάθουμε αυτά. Επανειλημμένα θα λέω. Το έχω ξαναπεί και νομίζω το συντομότερο θα πρέπει να μας ενημερώσετε. Τελευταίο, για τον Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Αν υπάρχει αίτημα αύξηση του προπολογισμού του, να το δούμε θετικά, αλλά να είναι δικαιολογημένο. Και θέλω να ακούσω ε, τεκμηρίωση, δικαιολόγηση, γιατί θέλουν περισσότερα θέματα. Δεν λέω να τα δώσουμε, αλλά ξέρουμε γιατί. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Όπως έλεγα, όταν έλαβα το λόγο. Είμαστε σε μια συγκυρία κρίσης. Και από ό,τι φαίνεται τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο θα κρατήσουν μια γραμμή λιτότητας. Αλλά έχουμε και τη θέση της συνθήκης της Λισαβόνας. Επομένως κινούμεθα σε ένα καινούριο πλαίσιο, καινούριο σκηνικό. Όμως ακόμα είναι νωρίς όσον αφορά την αποκριστάλωση αυτής της γνωμοδότησης για να δούμε τι θα προτείνουμε στην ε, Επιτροπή των Προπολογισμών για το χώρο δικαιοσύνης, ε, ελευθερίας κλπ. και ασφάλειας. Τέλος πάντων, για να ληφθεί κάποια απόφαση θέλουμε να γίνει μια και μόνη ανάγνωση για να συνοηθεί το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Ως συνομοθέτες. Το πλαίσιο της συναπόφασης και πρόκειται για ειδική διαδικασία εξαιρετικής φύσης. Μία και μόνη ανάγνωση λοιπόν. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνδιαλλαγή. Το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι αποδεικτό και από τα δύο θεσμικά όργανα. Η κυρία Βερζάτ. που είναι η σκιώδη συγγήτρια και ο κύριος Άλβαρο που είναι επίσης και ο θα πρέπει να βρεθούμε και να συνοηθούμε τόσο ώστε να καθορίσουμε ποιες είναι οι δικές μας προτεραιότητες. Γιατί ακριβώς αυτό εδώ είναι το θέμα. Να δούμε πώς και τι θα κάνουμε με αυτές τις, όλες αυτές τις προτάσεις, αυτές τις 14 δράσεις και καθώς και προγράμματα πιλωτικά για ασφάλεια δικαιοσύνη και να δούμε με ποιες προτεραιότητες θα μπορούσαμε να βρούμε την αναγκαία συνένεση. Για να μπορέσουμε να διεκπαιρώσουμε αυτό το θέμα. Πάρα πολύ βασικό το θέμα της θέσης ισχύης της Λισαβόνας. Άρα θα πρέπει τα δύσκολα τμήματα του προπολογισμού θα αφορούν την... τον έλεγχο ποιότητας Άρα θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο ακριβείς και προσεκτικοί για τα θέματα της εκτέλεσης του προπολογισμού. Για τις δαπάνες, δηλαδή. Τι θα γίνει, όπως είπαμε πολλές φορές, τι θα γίνει με τον έλεγχο των συνόρων. Τι θα γίνει με το SIS δεύτερη γενιά. Πάντω θέλω να σα πω ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο ελιγμών τον Ιούλιο τόσο ώστε να τα βρούμε με την Κομισιόν. Για να δούμε πού μπορεί να έχουμε αύξηση κονδυλίων τα οποία να βρουν το Συμβούλιο σύμφωνο. Μέσα σε αυτή την συγκυρία της χρηματοπιστωτικής χρήσης γιατί αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι ασφάλεια δικαιοσύνη και ε, ε, θα έχουν αύξηση πάνω από 2%. 12, 12, 12%. 12, 12. Και γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες θα έχουν αύξηση η οποία θα είναι ανάλογη με το τι ζητήσαν εκτός από την υπηρεσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι λεπτομέρειε του αιτήματο, αλλά έχει ένα λογικό αίτημα. Και ζητεί αύξηση 50% σε σχέση με πέρσι. Οπότε θα πρέπει εμείς να είμαστε ανοιχτή. Ε, μου ζήτησε ο διευθυντή τη υπηρεσία αυτή να συναντηθούμε για να τα συζητήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι λογικό να εγγράψουμε 50% 10 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από τα 10, από τα 20, από τα 20 που τους χορηγήθηκαν. Όμως Ας είμαστε ανοιχτοί για όλα αυτά τα παραπάνω που πάνε πέρα από το 5%. Να το εξετάσουμε και να δούμε σε ποια πλαίσια εντάσσεται αυτό το αίτημα της αύξησης για τον χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας. Άρα θα κάτσουμε να τα πούμε με τους σκιώδες Οπότε την επόμενη φορά θα συζητήσουμε τον Ιούλιο δηλαδή. Να κάτσουμε και να επεξεργαστούμε τις προτεραιότητές μας. Να δούμε πού μπορούμε να τα βρούμε. comments... Στα αγγλικά τώρα. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει κάτι να πει. Yes, the Commission. Ορίστε, Έχετε το λόγο. Ορίστε η Επιτροπή. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχει ένα θέμα. Ε, ναι, ναι, υπήρχε ένα ερώτημα που μου θέτει και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ερώτημα κυρίας Κούλερ για τη χρησιμοποίηση των κοντιλίων του Frontex. Μία εξήγηση είναι ότι οι καθυστερημένες αιτήσει των χωρών μελών για συνεισφορές από το Frontex. Υπάρχει κάποιος χρόνος που χρειάζεται για όλη τη διαδικασία και τα κράτη-μέλη συνήθως ζητούν την αποζημίωση καθυστερημένα. Και αυτό εξηγεί εν μέρη γιατί υπάρχουν πλεονάσματα. Τώρα, για τα signed revenue που λένε. Είναι ένας ε, δημοσιονομικός μηχανισμός αρκετά πολύπλοκος. Όταν ο κοινοτικός προϋπολογισμός χορηγεί κάτι, ένα κονδύλιο που δεν χρησιμοποιείται τελικά σε κάποια υπηρεσία, τότε ζητάει την επιστροφή του μη χρησιμοποιηθέντος τμήματος του κονδυλίου πάλι στον προϋπολογισμό αλλά το βάζει σε μια ειδική θέση του προϋπολογισμού. Τα ποσά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από το Frontex επανέρχονται στον προϋπολογισμό αλλά ξαναμπαίνουν για τον ίδιο σκοπό, για δράσεις Frontex δηλαδή, το επόμενο οικονομικό έτος. Αυτά είναι τα λεγόμενα προκαθορισμένα έσοδα. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι για την IT, για την ηλεκτρονική, τα περισσότερα ποσά έχουν μπει στο αποθεματικό δηλαδή. Αν όλα γίνουν κανονικά, από το 2011 και μετά θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να προσλαμβάνουμε κόσμο. Και γι' αυτό ζητήσαμε τα κονδύλια, αλλά είναι προς το παρόν στο απόθεμα μέχρι να καθοριστεί πλήρως η λειτουργία της υπηρεσίας αυτής. Της ηλεκτρονικής. Τώρα το αίτημα του κυρίου Μπουσουτήλ για την αναθεώρηση της εντολής του Frontex. Η είχε θελήσει να επιδείξει κάποια φρόνηση για τον προϋπολογισμό του Frontex, πράγμα που ισχύει για όλες τις υπηρεσίες. Θελήσαμε να βασιστούμε στην πραγματική χρήση των θέσεων του προϋπολογισμού και των προγραμμάτων των προηγουμένων ετών και βέβαια είμαστε διατεθειμένοι να ζητήσουμε και πρόσθετα κονδύλια εάν μας υποβληθούν συγκεκριμένα προγράμματα όπως για την αγορά εγκαταστάσεων ή υλικού που προς στιγμή δεν έχει γίνει. Για τα ταμεία μία μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση θα γίνει το φθινόπωρο. Σας υπενθυμίζω ότι τα προγράμματα αυτά άρχισαν να ισχύουν το 7 με κάποια καθυστέρηση γιατί καθυστέρησε η έγκριση της νομικής τους βάσης και στην ουσία δεν άρχισαν πριν το 8. Η δε μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση θα γίνει το Φεβρουάριο, κατά τα τέλη του έτους δηλαδή. Το φθινόπωρο με συγχωρείτε. Να, αυτά σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν συμφωνείτε λοιπόν, κύριε Βαντεκάμπ, θα μπορούσαμε να συγκαλέσουμε ε, συνεδρίαση των συντονιστών ε, στο Στρασβούργο στην επόμενη σύνοδο για να συναντηθούμε ο κύριος Βαντεκάμπ, η κυρία Βερζάτ, η ο κύριος Άλβαρο και να πούμε σε λεπτομέρειες, έτσι για να μπορέσουμε να δώσουμε γνωμοδότηση τελικά με την οποία να μπορούν να συμφωνήσουν οι πολιτικές ομάδες, να τους ικανοποιεί δηλαδή. και να στείλει και πολιτικό μήνυμα από την Επιτροπή Ελευθεριών στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συμφωνείτε έτσι. Ορίστε κύριε Βαντακάμπ. Ναι, μια παρατήρηση μόνο αν μου επιτρέπετε. Συμφωνώ με την κυρία Κέλλερ και προηγουμένως πριν να έρθουμε σε επαφή με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για να ξέρουμε ποιες είναι πραγματικές τους ανάγκες πριν γίνει αυτή η συνεδρίαση. Καν. Of course, I made that... Ναι, βεβαίως, το είπα και εγώ. Έχω λάβει ενημέρωση ε, από το ε, οργανισμό αυτό και ζητούν ούτε λίγο ούτε πολύ 50% αύξηση χρηματοδότησης. Ε, θα πρέπει να δούμε γιατί ε, τα ζητούν αυτά. Είναι αιτιολογημένα, είναι λογικά. Γιατί αύξησε κατά 50%. Είναι εφικτά, είναι σωστά και γίνεται και σε τέτοιους καιρούς δημοσιονομικούς που ζούμε. Όλα αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξουμε. Να κανονίσουμε ε, να κανονίσουμε συνάντηση με τον Διευθυντή, ο οποίος ζήτησε ειδικά συνάντηση μαζί μας και με τους συντονιστές και τα μέλη της Επιτροπής για να έχουμε και η ε, ε, άποψη, η ιδέα για ποιους λόγους ζητούν τόσα πολλά χρήματα. Εντάξει. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Φτάνει για σήμερα ε, στην προγραμματισμένη ημερησία διάταξη για την απογευματινή συνεδρίαση. Όσοι δεν είναι συντονιστές και δεν μπορούν να συμμετέχουν, έχουμε και κλεισμένο το θυρών συνεδρίαση, παρακαλούνται να αποχωρήσουν. Είναι και κλεισμένο το θυρών συνεδρίαση των συντονιστών. Απουσιάζουν όμως, δεν βλέπω τον κύριο Άλβαρο, ούτε τον κύριο Μωράες, που είναι συντονιστές. Θα τους τηλεφωνήσουμε. Το συντομότερο να αρχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι υπόλοιποι αύριο το πρωί στις 9 γιατί θα έρθει ο Υπουργός, δύο Υπουργοί, Ισπανική Προεδρία, Υπουργό ε, Ρουμπαλκάμπα Εσωτερικών και ο Υπουργό Καμάνιο Δικαιοσύνης, στις 9 η ώρα ακριβώ.